διεξήχθησαν εκεί και θέλω να τονίσω δύο πράγματα, δύο θέματα, τα οποία είδα εκεί. Αφενός τον ρόλο του IGF, εφόσον παραμείνει αυτή η πολυμερή συζήτηση μεταξύ πολλών stakeholder, το άλλο, το θέμα της διακυβέρνησης του διαδικτύου. διεξήχθη συζήτηση σε διάφορες συνεδριάσεις, αλλά μιλήσαμε και με άλλους εκεί για το αν θα διατηρήσουμε το IGF όπως είναι τώρα, συζήτηση δηλαδή μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, συζήτηση χωρίς τελική θέση και από την άλλη μεριά, το δεύτερο θέμα, είναι της διάσκεψης στην Βραζιλία, όπου η βραζιλιάνικη κυβέρνηση πιθανώς θέλει να προχωρήσει σε επανακαθορισμό της διακυβέρνησης του διαδικτύου. Σκοπεύει να οργανώσει την συνεδρία σε αυτή το 2014. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το τι θα συζητηθεί. Ούτε πώς θα γίνει η οργάνωση, ούτε ποιοι θα συμμετέχουν. Αλλά πάντως είναι ευκαιρία για να οριστούν ξανά οι ρόλοι της, ε, ο ρόλος μάλλον της κυβέρνησης του δικτύου στο μέλλον. Και ένα σχόλιο για μια από τις ε, συναντήσεις, πολύ σημαντική για μένα, με τον CEO της ICAN, που όταν συζητήσαμε για το θέμα αυτό, για τη Βραζιλία και το μέλλον της ε, διακυβέρνησης του διαδικτύου, Είναι καλά, εξηγείται καλά και στην έκθεση της γραμματείας, αλλά εξήγησε πώς έχει αναπτυχθεί το ΙΚΑΝ μέχρι τώρα, αλλά η συζήτηση που γίνεται είναι και αν θα πρέπει το ΙΚΑΝ να εξαρτάται ακόμη από τον νόμο της Καλιφόρνιας, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή, ή αν θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα πιο διεθνές πλαίσιο. είπε ότι είναι δυνατόν αυτό, να υπάρξει πιο διεθνής διακυβέρνηση του ΕΚΑΝ αλλά μας είπε επίσης ότι η κυβέρνηση των Ενωμένων Πολιτειών είναι, είναι έτοιμη να προχωρήσει, αλλά ότι πρέπει να έχουμε υπόψη και την ανάγκη να διατηρηθεί το καθεστώς του ίντερνετ και η ισχύς του και ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το μοντέλο αν δεν είμαστε σε θέση να ορίσουμε ένα καινούριο μοντέλο. Και αυτό πιθανότατα θα τεθεί επιτάπητος και στην Βραζιλία. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρετηθούν του ελέγχου του διαδικτύου υπέρ κάποιου άλλου οργανισμού, αν δεν ξέρουν πώς θα λειτουργεί αυτός ο οργανισμός. Αυτό είπε ο διευθυντής του ΕΚΑΝ με αυτό μας είπε δηλαδή. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος που θέλει να θέσει ερωτήσεις? Όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους ε, για την ενημέρωση σχετικά με την αποστολή. Τώρα θα διακόψουμε τις εργασίες μας ε, μέχρι τις 4 για να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ε, καθές, όπως ξέρετε, είναι καθορισμένη η ώρα των ψηφοφοριών. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στις 4.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 Cari colleghi, possiamo Να ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι με τις ψηφοφορίες. Θα σας παρακαλούσα να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία καταρχήν. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίστε σας παρακαλώ για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Avete votato tutti? Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Όχι. Παρακαλώ. Κύριε Μπουτικόφερ. Κύριε Πρόεδρε, ξέχασα την κάρτα μου. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε κάτι παρατρίχα, να, να είναι η ψηφοφορία κοντά-κοντά, θα κάνω ένα νόημα. Θα σας παρατηρεί η γραμματεία. Και εγώ το ίδιο, μάλιστα δύο. Ευτυχώς είστε από την ίδια ομάδα, μας διευκολύνει. Μάλιστα, ωραία. Ξεκινάμε με την έκθεση σαρτόρι, Συμβασμός με το Συμβούλιο. Υπέρ. Ηλεκτρονικά πρέπει να ψηφίσουμε, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 31. 31 ψήφι περ, μία κατά και δύο αποχές. Ας περάσουμε στη δεύτερη έκθεση Σαρτόρη για τη Συμφωνία Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Τρει-πέντε υπέρ και μία ψήφος κατά. Ωραία. Περνάμε τώρα στην έκθεση Duke. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Έλεγχο για το 9. 39. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2. Υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά απόχέ, συγκρίνεται 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά απόχέ, συγκρίνεται 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές ρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 και 22 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 και 25 μαζί υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, παρακαλώ, έλεγχος για την 67 παρακαλώ. Πέρας. 20 υπέρ και κατά. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 70. Συγγνώμη, 50 διορθώνει η πρόεδρος. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 και 21 μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 83 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ, κατά, εποχέ, απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά, εποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά, εποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Τροπολογία 8 ίντα. Σας βλέπω κάπως ε, χαμένους. Μετάδοση συμβαστική 5. Δεν το ψηφίζουμε, περνάμε στην 101. Ένα λεπτό για να είμαστε σίγουροι. να κάνουμε μια παλήθευση. Τι λέει ο εισηγητής, πρέπει να ψηφίσουμε ή όχι on va les voter, mais plus tard. Eh Μου λέει η γραμματεία ότι θα ψηφίσουμε αργότερα την τροπολογία 8. 101 λοιπόν. Τροπολογία 101. Έτοιμοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά σε παληθεύσουμε. Δεν βλάπτει για την 101. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. 26 υπέρ 12 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 130. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 108. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 110. Υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 113. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114. Υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 115. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 116. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 138 σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9 ναι. υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Όχι. Τροπολογία 6 υπέρ Αν ο συμβεσμός 9 υιοθετήθηκε, επομένως, καταπίπτει συμβαστική 12. Επομένως, περνάμε απευθεία στην τροπολογία 6. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για την 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τριάντα υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 145 και 7 μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. γιατί είναι 146 απορρίπτεται. Τώρα 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 148. Και είναι τα 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβασμός 10. Υπέρ, κατά. Εποχές εγκρίνεται. Το πίπτη. Συμβιβαστική 13. Και πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 8 από πριν. Είναι τα 8 που δεν την ψηφίσαμε προηγουμένως. Εντάξει, υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται, Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται, Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 152. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 153. Έλεγχος για την 152. Άρχεται ψηφοφορία. πέρα. 5 υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 172 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 170 τα υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά εδώ με μπερδέψατε τροπολογία 10 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14, Περ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 20, Περ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 την 23 Μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 23. Μας ζήτησαν να επαληθεύσουμε την τροπολογία 23. Πέρας. 26 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται.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 απολύπτονται. Τροπολογία 2 και τροπολογία 1 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τη Της απασχόληση Απασχόληση Υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 30 υπέρ, 5 κατά, 7 και 4 εποχές. Τώρα περνάμε στην έκθεση Anders Dotter. Έτοιμοι. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 59 παρακαλώ. Πέρας. 10 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άφετ 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει ένα αίτημα από τον συνάδελφο Πρόντι να ψηφίσουμε την τροπολογία 76 πρόσθετα, πρόσθετη ψηφορία υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 77. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Πέντε υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται. Άφετε 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78. Τικάου. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι πρώτη πέρα κατά αποχές απορρίπτεται άφετ 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 19 υπέρ κατά απόχε εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 και 82 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτω. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Budget 5 και 83 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 21, 36, 9, 10, 55, όλες μαζί υπέρ, κατά εποχές εγκρίνονται. 86 υπέρ, κατά εποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Συμβιβασμός 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 26 και 27 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άβετ 28 υπέρ. Κατά εποχές γκριντ. 99, 49, 50 και 52 μαζί. Υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές γκριντ. Συμβαστική 14 και συμβαστική 7 σε μπλοκ μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τα καλό. Ψηφίσαμε το συμβασμό 14 και το συμβασμό 7 μαζί γιατί υπάρχει διαφορετική αρρύθμιση στις σελίδες. Το βρήκατε. Πολύ ωραία. Πάμε στην budget 8. 8, 9, 13 και 3. Υπέρ, κατά. Εποχές συγκρίνονται. 108 και 11 μαζί. Υπέρ. 108 και 11 σε μπλοκ. Υπέρ. Κατά. Να κάνουμε μια επαλήθευση για τις τροπολογίες 108 και 11 μαζί. Πέρας. 20 υπέρ, 19 κατά. 22 υπέρ. Απορρίπτεται. Οι δύο βέρδι δεν έχουν la τέσσερα, no? Οι δύο πράσινοι δεν έχουν την κάρτα. Συνάδελφοι Μπουτικόφερ και Λάμπερτ. Τροπολογία 109. Υπέρ. Και 9 πρώτη, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άφετ 30, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άφετ 31, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άφετ 32, υπέρ, Κατά. εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άφετα 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 6 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται 7 κατά εποχές, εγκρίνεται τροπολογία 44 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται αφετ 8 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφετ 9 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τώρα έχουμε τις ψηφορίες για τις τροπολογίες. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Σαράντα μία ψηφέρ, μία κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο συνολό του, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 49. εγκρίνεται. Και έχουμε τώρα την ε, ψηφοφορία για τις διαπραγματεύσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Σε υπέρ, μία κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση Πιλάρ Δελκαστήγιο. Έτοιμοι. Τροπολογία 26 πέρα. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 203 πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 204D. Υπέρ. Κατά. σε απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη 206. έλεγχος. Πέρας. 20 υπέρ, 20 κατά. Είκοσι υπέρ και 21 κατά. Απορρίπτεται. 207. Υπέρ κατά. Χες. Απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές, συγγνώμη, 211 και 212 μαζί, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 213 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 214 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 και 215 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29D και 216D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 224 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 225 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 32, 33, 34 μαζί υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 226 και 228 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 227 Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 229. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 230. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 231. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 233. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 234 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 235 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 39 και 40 μαζί υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 236 υπέρ κατά αποχές 46 Σαράντα 238-239 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 242 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 243 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 265 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 268 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογή 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 282 έλεγχος. Έλεγχος. Είναι το 282. Πέρας. Απορρίπτεται. 283. Περ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 285. Περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 287. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 71 και 288 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 310 και εδώ έχουμε έτοιμη προφορικής τροπολογίας ε, από τη συνάδελφο Χέλλερ. Θέλετε να το παρουσιάσετε και να δούμε αν το δέχονται οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Η τροπολογία αυτή... Σε εθελούσια βάση θέλουμε οι φορείς της αγοράς να ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς για ενδεχόμενες απώλειες και είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και ε, των Αμερικανών και τα δικά μας. Τώρα, ε, σε θελοντική βάση, το FCC ζητά από τις Αμερικανικές εταιρείες να το κάνουν και επαναλαμβάνω γίνεται πάντα σε εθελοντική βάση. Στα πλαίσια του διατλαντικού νομοθετικού διαλόγου θέλουμε να έχουμε σε κάποιο βαθμό μία εναρμόνιση της νομοθεσίας και γι' αυτό είχαμε σκοπό να το προσθέσουμε εδώ. Σήμερα λοιπόν συμφωνήσαμε με τους ελιστές και τους πράσινους ότι για το ε, το incident, δηλαδή το επεισόδιο, το, το, το αλλάζουμε και το κάνουμε απώλειες, οικονομικές απώλειες. Οπότε για τις οικονομικές απώλειες δεν χρειάζεται να δοθεί κάποια εξήγηση, απλώς μια ενημέρωση, δεν χρειάζεται δηλαδή μια περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Δηλαδή μια τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσει για το αν κάποιος τη λίστεψε. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει αν έχει χάσει κάποια χρήματα μέσω κάποιας κυβερνοεπίθεσης. Άρα λοιπόν είναι σε θελοντική βάση και είναι μία ενημέρωση ε, για απώλεια οικονομική αντίστοιχη με αυτό που γίνεται σε θελοντική βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιλάρ Η κυρία Δεν πρόκειται να σας εξηγήσω για ποιο λόγο η θέση μου είναι να ψηφίσουμε κατά θα σας ε, πω στους συναδέλφους του ΕΛ και στους υπόλοιπους πως εγώ αυτή τη στιγμή διατηρώ την αρνητική θέση που έχω για αυτή την αλλαγή. Βάζω λοιπόν ένα πλήν. Συμφωνείτε όλοι με την προφορική τροπολογία. Φαίνεται να γίνεται αποδεκτή. Συμφωνούν όλοι με την προφορική τροπολογία, όχι? Παρακαλώ. Δεν συμφωνεί η ομάδα μου. συμφωνεί ομάδα μου για αυτή την προφορική τροπολογία. Δεν θα ψηφίσουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία. Θα ψηφίσουμε μόνο την 310 χωρίς την προφορική τροπολογία από την κόφερ. Παρακαλώ. Εγώ πληροφορήθηκα ότι η προφορική αυτή τροποποίηση έγινε για ένα και μόνο λόγο. Λόγω συμβιβασμού με τον σκιώδη εισηγητή της σοσιαλιστικής ομάδος, κύριο Κάλφιν. Δεν κατανοώ λοιπόν για ποιο λόγο τώρα λέγουν οι σοσιαλιστές ότι δεν την υποστηρίζουν. Αυτά δηλαδή που εμείς έχουμε συμφωνήσει ως παραχώρηση απέναντι στους σκιώδη ηγητή τους. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω φυσικά γι' αυτό. Εγώ ξέρω μόνο ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή η προφορική τροπολογία, αρκεί τρεις-τέσσερις να μην είναι σύμφωνοι και δεν γίνεται δεκτή η προφορική τροπολογία. Θα ήθελα ε, να με συγχωρήστε για τη σύγχυση, δεχόμαστε την προφορική τροπολογία, αλλά θα την καταψηφίσουμε, αυτό είπα. Eh, Μάλιστα, δηλαδή δεν υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία, οπότε θα ψηφίσουμε μαζί με την 310, άρχεται ψηφοφορία. Ο κύριος Τσίτσεστερ. Uh, Λυπάμαι κυρία Πρόεδρε, αλλά είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας. Οπότε δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Ποιο ε Ποιος είναι κατά της προφορικής τροπολογίας. Χρειάζονται τέσσερα άτομα για να απορριφθεί. Μάλιστα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία 310 ως έχει. Άρχεται η ψηφοφορία. Και έτσι δεν θα έχουμε και προβλήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 335 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 337 υπέρ. Κατά εποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 336 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 338 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 342 υπέρ. ...342, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 343, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 96, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 344 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 345 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κα... Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 143 με προφορική τροπολογία του κ. Τσουκαλά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144. 145 με συγχωρείτε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 περ κατά αποχές εγκρίνεται 171 περ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 182 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, απόχε εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά αποχέ συγκρίνεται, 21 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά απόχε, συγκρίνεται, 201 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πέρας. δεύτερα υπέρ. Έξι κατά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην συγγήτρια. Adesso noi eh, abbiamo il TNT, prima di tutto... Λοιπόν, τώρα, να ξεκινήσουμε τώρα με το ψήφισμα και κατόπιν θα περάσουμε στην ε, προφορική ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε με το ψήφισμα για την έκθεση Ρούμπι. Παρακαλώ, συμφωνείτε. Το ψήφισμα. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εποχέ συγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτει. 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτει. Έλεγχο για τη 14 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Πέρα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 20, υπέρ, κατά αποχές γκρίνεται, 21 σε δύο μέρη, πρώτο μέρος υπέρ, κατά αποχές γκρίνεται, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές γκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ, κατά αποχές γκρίνεται. Συμβασμός 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. Συμβασμό 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για τον συμβιβασμό 5 έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 25 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 32, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41, 42 διορθώνει πρόεδρος, τροπολογία 42, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για τις 44. Πέρας. 25 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται.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 κατά αποχές αγκρίνεται, τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές αγκρίνεται, τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές αγκρίνεται, 5 υπέρ, κατά αποχές αγκρίνεται, 6 υπέρ, κατά αποχές αγκρίνεται, 7 υπέρ, κατά αποχές αγκρίνεται, 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, άρχεται ψηφοφορία. Votazione. Πέρας. 26 υπέρ, 14 κατά, 17 κατά και μία εποχή. Εγκρίθηκε λοιπόν το ψήφισμα και περνάμε τώρα στην προφορική ερώτηση για το top 10, Rubik και πάλι, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Πέρας. τέσσερις υπέρ, 4 κατά, 5 εποχές. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Να διακόψουμε για 3 λεπτά όποιον θέλει να αποχωρήσει. Και θα συνεχίσουμε με τις εργασίες της Επιτροπής.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 que nous avons On a encore Madame, Madame Jordan et après, après Madame Corolla. Bene, proseguiamo i nostri lavori. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας με την έκθεση της κυρίας Τζόρνταν και της δίνω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Πρέγω, Ρωμάνα. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ. Το Μάρτιο του 2011, ε, του 12 με συγχωρείτε, είχαμε την καταστροφή στην Φουκοσίμα. Τότε λήφθηκε μία απόφαση να γίνει μία σειρά ε, δοκιμών αντοχής στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης και βάσει αυτών των ε, δοκιμών να γίνει μία αναθεώρηση της τρέχουσας νομοθεσίας για την, για την πυρηνική ασφάλεια. Αυτό κάναμε και έχουμε μπροστά μας μία πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, μελλοντική οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια και έχουμε και κάποιες τροπολογίες. Έχουμε αρκετές νέες εξελίξεις, αρκετές τροπολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη γνώμη μου, έκανε πολύ καλή δουλειά και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις προτάσεις που γίνονται. Ε, Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξέτασε προσεκτικά τον ορισμό. Δηλαδή ποια είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Επίσης, η πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνει και κάποια κριτήρια για το τι ακριβώς, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος αυτής της ε, ε, αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, ε, πώς θα πρέπει να περιγράφεται αυτή και θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος φορέας και επίσης θα πρέπει να είναι οργανωμένη με συγκεκριμένο τρόπο, να έχει περικοδοτείται με επαρκή προϋπολογισμό, να έχει νομικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες και το κατάλληλο ε, ανθρώπινο δυναμικό και πόρους. Επίσης, θα πρέπει να ε, επιβλέπει το θέμα της απόκρισης σε επίγουσες καταστάσεις, κάτι το οποίο περιγράφεται και με περισσότερες λεπτομέρειες στο διατακτικό. Επίσης, στην πρόταση αυτή έχει συμπεριληφθεί μία σειρά άρθρων για τους κατόχους των αδειών. Εδώ έχουμε και πάλι έναν επανακαθορισμό ε, του τι σημαίνει peer review. Και εδώ επίσης αναφέρονται οι ανθρώπινοι πόροι με μεγαλύτερες λεπτομέρειες, δηλαδή όσοι θα κάνουν αυτό το peer review θα πρέπει να έχουν τις δεξιότητες ε, και τις γνώσεις για να κάνουν αυτή την αξιολόγηση. Και έχουμε και μία νέα υποχρέωση για την καταλληλότητα την οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν και να τεκμηριώνουν οι υπεργολάβοι. Επίσης, το θέμα της διαφάνειας. Και εδώ, επίσης, έχουμε μια νέα απέτηση για την Εθνική Αρμόδια Αρχή, όπως επίσης και για τον φορέα και τον κάτοχο της αδειοδότησης, να χαράξουν μια ε, ικανοποιητική στρατηγική για τη διαφάνεια. Έχουμε να συμπεριλάβει και ένα κεφάλαιο για τις ειδικέ υποχρεώσεις, δηλαδή ποιοι είναι οι στόχοι γενικής ασφάλειας και πώς θα εφαρμοστούν η μεθοδολογία. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν αυτή η νομοθετική πρόταση συμπεριλαμβάνει πολύ σημαντικές ε, προτάσεις για το πώς κανείς μπορεί να εφαρμόσει ε, την ε, ε, κουλτούρα ασφάλειας που επιβάλλεται και θα πρέπει οι στόχοι ασφάλειας να καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των πυρηνικών εγκαταστάσεων, δηλαδή από τη στιγμή της χωροθέτησης, της οικοδόμησης, μέχρι λοιπόν και ε, του παροπλισμού αυτών των εγκαταστάσεων. Από αυτές τις ε, πρόσφατες ε, καταστροφές έχουμε διδαχθεί πολλά. Μπορούμε να δούμε ποιοι είναι οι εξωτερικοί κίνδυνοι οι οποίοι μας απειλούν και ποιοι είναι ε, οι, εξωτερικοί κίνδυνοι που προέρχονται όχι μόνο από τη φύση αλλά και από την ανθρώπινη δράση. Κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι πως διάφορων, διαφορών ειδών καταστροφές συμπεριλαμβάνονται εδώ. Το κείμενο λοιπόν είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Αναφέρεται δηλαδή στην οικοδόμηση ε, και στην, ε, στα προβλήματα που μπορεί να ε, προκαλέσει η λανθασμένη κατασκευή, ο λανθασμένος σχεδιασμός και αναφέρεται και στα ατυχήματα με βαθμό σοβαρότητας. Επίσης, τι συμβαίνει αν έχει πληγεί ο πυρήνας στον αντιδραστήρα, γίνονται λεπτομερείς αναφορές και το γεγονός πως δεν θα πρέπει οποιαδήποτε καταστροφή να ξεφύγει από την περιοχή περιορισμού. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να είναι κανείς πάντα έτοιμος και να υπάρχει μια απόκριση στις ίδιες, μια πρώτη απόκριση ήδη on-site στις εγκαταστάσεις ο σχεδιασμός να έχει προβλέψει τέτοιου είδους προβλήματα και αυτό το οποίο διδαχθήκαμε από την Ιαπωνία είναι πως είναι πολύ σημαντικό αυτές οι πυρηνικές εγκαταστάσεις να έχουν μια κεντρική μονάδα η οποία θα προστατεύεται παρκώς από φυσικές καταστροφές. Αν δηλαδή συμβεί οτιδήποτε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε με τη λειτουργία ολόκληρης εγκατάστασης από κάποια κεντρική μονάδα. Επίσης έχουμε νέες απαιτήσει για το peer review, έχουμε αυτές τις ε, αναδεκαετία τακτικές ε, αναθεωρήσεις και εξετάσεις όπως επίσης και τις εξαετήσει που γίνονται σε θεματικό επίπεδο. Ως τμήμα λοιπόν αυτών των αξιολογήσεων ενισχύεται και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι θετικό. Αυτό επίσης αποτελεί ένα από τα μαθήματα της Ιαπωνίας. Εκεί ήταν εξαιρετικά αποδυναμωμένη η ρυθμιστική αρχή και δεν βρέθηκε κανείς να αποκαλύψει το κακό κείμενα. Νομίζω ότι εμείς εδώ δίνουμε την προστιθέμενη αξία την οποία προσφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το επίπεδο. Κυρώσεις τώρα, ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, να σας πω στα γρήγορα τι συμβαίνει. Εμείς περιμένουμε τις τροπολογίες αυτές, τις τροποποιήσεις στην οδηγία για την ασφάλεια και νομίζω έφτασαν την κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε να εγκριθούν μέχρι το τέλος της θητείας, αλλά θα πρέπει να πιεστούμε, να σας πω πως οι δικοί μου συνεργάτες εργάζονται σκληρά και στόχος μας είναι να είναι η έκθεση έτοιμη μέχρι αύριο έτσι ώστε να υποβληθεί για μετάφραση και μετά στην πρώτη ολομέλεια του Απριλίου να ψηφίσουμε. Επίσης σχεδιάζουμε και μια ακρόαση για τις 12 Φεβρουαρίου. Επί της ουσίας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα θα ήθελα να μειωθεί στο μέγιστο αριθμό των διαφόρων επεισοδίων ή ατυχημάτων, αλλά ό,τι και να κάνει κανείς, πάντα υπάρχει η πιθανότητα κάτι τέτοιο να συμβεί. Οπότε χρειάζεται να είμαστε πάντα ε, έτοιμοι να μπορούμε να δώσουμε μια γρήγορη απόκριση και καλό συντονισμό. Θα ήθελα να είναι πιο ενιαίοι οι κανόνε που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα βελτίωνε και τον τρόπο με τον οποίο μα αντιμετωπίζουν οι πολίτε, γι' αυτό τον τύπο ενέργεια, να τον εμπιστεύονται περισσότερο και γι' αυτό η εξαετή θεματική αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω ένα κίνητρο για περαιτέρω εναρμόνιση. Όπω είπατε και εσεί, οι προτάσει τι οποίε κατέθεσε ο Επίτροπο είναι σωστέ και νομίζω ότι με αυτά τα σχόλια που έκανα, που ήταν επί τη ουσία, ε, και με κάποιες τεχνικές τροπολογίες, στις οποίες πιστεύω πως θα πρέπει ε, να ακολουθήσουμε περισσότερο τις, ε, τα πρότυπα της Διεθνούς Αρχής Ενέργειας, να καταφέρουμε ένα πολύ ευνοϊκό για μας κείμενο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορέιδα παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γενικά, Συμφωνώ με την συγκήτρια. Το περίτεστατικό, το τύχημα της Κοσίμα έχει οδηγήσει την κοινή γνώμη να ανησυχεί για το τι συμβαίνει και αποκαλύπτει και την ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων πολύ σοβαρών και κατόπιν του ατυχήματο ε, λήφθησαν ε, πάρα πολλές αποφάσεις, πολύ σημαντικέ ε, για το θέμα του μέλλοντο τη πυρηνικη ενεργειας ενέργειας. Διάφορα κράτη-μέλη έλαβαν αποκλίνουσες θέσεις, όμως η πυρηνική ασφάλεια δεν έχει σύνορα και η αλήθεια είναι ότι είναι διασυνορική ακόμη και ενδιαφέρουν οι πολιτικές των κρατών μελών. Γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε τα επίπεδα ασφαλείας στην ευρωπαϊκή επικράτεια όπου συγκεντρώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο το 1 τρίτο των πυρηνικών αντιδραστήρων σε λειτουργία. θεώρηση τώρα της νομοθεσίας και η ανάλυση είναι ευπρόσδεκτες και θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε και τα διδάγματα του ατυχήματο Φουκουσίμα και των stress test που έγιναν στι πυρηνικέ εγκαταστάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να ενισχύσουμε την εξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, τη διαφάνεια, την ικανότητα των μηχανισμών συντονισμού και συνεργασία μεταξύ αυτών των εντοτήτων και ιδίω μέσω μηχανισμών αξιολόγηση ομοτήμων την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ουσιαστική για την ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας. Η πρόταση σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, όμως επίσης ενισχύει το ρυθμιστικό ρόλο της Κομισιόν καθορίζει αρχές και δίνει προσανατολισμούς για δομές και διαδικασίες ασφαλείας που να αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές. Πρέπει οι στόχοι ασφάλειας σε ψηλό επίπεδο να καλύπτουν τα διάφορα στάδια του κύκλου της ζωής των πυρηνικών εγκαταστάσεων από την επιλογή της τοποθεσίας μέχρι τον προπλισμό τους. Επίσης, είναι πρόσδεκτες οι προτάσεις για τις τεχνικές διατάξεις προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία και αποτελεσματική και ταχεία απάντηση σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Και γι' αυτό είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους σε αυτό το φάκελο και συγκεκριμένα με την εισηγήτρια και γενικά συμφωνούμε με τα συμπεράσματά της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο <clears throat> Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, τα είπαν τα πιο πολλά οι συναδελφοί μου, μετά από το ατύχημα της Φουκουσίμα, αυτό το τεραστίων διαστάσεων ατύχημα, βεβαίως το κοινό έχει ανησυχήσει πολύ. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και γι' αυτό έχουν γίνει πολλές δοκιμασίες που είχαν στόχο να εξετάσουν κατά πόσο είναι ασφαλή οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Βέβαια και θέλουμε να εναρμονίσουμε τον χώρο, να βελτιώσουμε την εναρμόνιση και ιδίως να ενισχύσουμε τον ανεξάρτητο χαρακτήρα των εθνικών εποπτικών οργάνων και να εξασφαλίσουμε διαφάνεια στην διαδικασία. Πολύ θετικό αυτό, διότι αυτό που θέλουμε είναι να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία στα μάτια του κοινού των περίπλοκων αυτών εγκαταστάσεων. Η τελική έκθεση της ΕΝΣΕΚ που διεξήγαγε αυτές τις δοκιμασίες αντοχής εντοπίζει τέσσερις τομείς βελτιώσεως ελέγχων αλλά δεν περιέλαβαν πρόταση για νέα βαθύτερη αναθεώρηση. Και αυτό νομίζω ότι αποτελεί πρόβλημα. Γιατί χρειαζόμαστε νέους ορισμούς. Πρέπει τα πράγματα αυτά να είναι πολύ καθαρά ορισμένα, έτσι ώστε να μην μένουν χώροι για παρανοήσεις. Και όταν μιλούμε για τους ελέγχους, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή. Για να μην υπάρξει απολύτως καμία, κανένα περιθώριο παρελμηνίας ώστε όλοι να γνωρίζουν, όλοι οι οργανισμοί να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά που ε, έγκυται τα καθήκοντά τους. Αυτό το νέο άρθρο 8α που προβλέπει την εξέταση από ομοτήμους πρέπει να εξηγηθεί πολύ καλά, διότι θεωρώ ότι δεν είναι απόλυτα σαφές το περιεχόμενο. Εάν έχουμε δύο διαφορετικές διαδικασίες μηχανισμών ελέγχου, ποιος θα αξιολογήσει ποιος είναι καλύτερος, ποιος μηχανισμός ελέγχου είναι καλύτερος. Γι' αυτό η πρόταση της Κομισιόν πρέπει να καταργήσει τις περιτές αυτές άλλωστε γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Διότι όλα αυτά είναι δυσκίνητοι μηχανισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε επιβράδυνση. Γι' αυτό και είναι σαφές ότι πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρος ο ρόλος των ρυθμιστικών οργάνων. Πιστεύω λοιπόν ότι ο οργανισμός που συνέταξε αυτά είναι βέβαιος επαγγελματικό και θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις δικές τους προτάσεις. Για το άρθρο 8 που μίλησα πριν, ορίζει και ποιος είναι ο ανεξάρτητος χαρακτήρας και αν η Κομισιόν θέλει να εποπτεύει, μπορεί τότε να σημειωθεί ενδεχομένως σύγκρουση συμφερόντων, γιατί η Κομισιόν είναι σε λίγο διαφορετική θέση. Γι' αυτό πιστεύω ότι το έγγραφο ως έχει υποβληθεί πρέπει να ξεκαθαρίζει τις επιμέρους αρμοδιότητες. Τι σημαίνει τι σημαίνει ο χώρος της ε, αρμοδιότητας, του ελέγχου κτλ. και ποια διαδικαστικά βήματα λαμβάνονται. Εγώ θα προτείνω να διεξαχθεί ακρόαση για το θέμα. Το βρίσκω πολύ σημαντικό γιατί μιλούμε εδώ για πολύ σημαντικές διαδικασίες που άπτονται τεχνικών, των τεχνικών πτυχών αυτών των πολύ περίπλοκων εγκαταστάσεων. Και επομένω αυτά πρέπει να μπουν σε λεπτομέρειε. Συζητήσει πρέπει να μπουν σε λεπτομέρειε. Εγώ πολύ ευχαρίστω να συνεργαστώ με την εισηγήτρια για το περίπλοκο αυτό θέμα. Να συνεργαστούμε στενά. Και όπω είπα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Από την άλλη μεριά, να μην υποκύψουμε στο ψυχολογικό βάρος και στις αμφολίες που εκφράζει το κοινό. Γιατί ξαναλέγω, μιλούμε για πολύ τεχνικού χαρακτήρα περίπλοκες εγκαταστάσεις και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο. Ευχαρίστως λοιπόν να συνεργαστώ με κάθε τρόπο στο έργο της. Η Επιτροπή, εφόσον επιθυμεί να βαρέμβει. Κυρία Συγήτρια, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα θερμά λόγια που μας απευθύνατε. Να σας υπενθυμίσω κάποιες κομβικές αρχές της πρότασής μας και θα ήθελα με τον τρόπο αυτό να εξηγήσω από πού προέρχονται αυτές οι προτάσεις, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τα όσα είπε ο προλαλής σας. Εμείς λάβαμε μια διπλή εντολή το 2011 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα δοκιμές αντοχής και δεύτερον αναθεώρηση και ενδεχομένως τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την πυρηνική ασφάλεια εφόσον χρειάζεται. Έχουμε λοιπόν το ψήφισμα το οποίο έχει καλέσει, μας έχει καλέσει να αναθεωρήσουμε την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια. Εμείς Συνεργαστήκαμε με αρκετές ε, οργανώσεις, όπως για παράδειγμα διεθνής, ε, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, τους εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές και συνεργαστήκαμε επίσης και με το κοινό μέσω των ακροάσεων που οργανώσαμε κατά τη διάρκεια των δοκιμών αντοχής. Εμείς Κάναμε επίσης ε, και κάποιες διαβουλεύσεις με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων, όπως κάναμε για την αναθεώρηση της Euratom. Όλα αυτά λοιπόν είναι αρκετά σφαιρικά και βασίζεται σε μια σειρά αρχών. Πρώτα απ' όλα, η ανεξαρτησία ε, των όσων παίρνουν τις αποφάσεις για θέματα ασφάλειας. Δεύτερον, η διαφάνεια της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων. τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας με την σύσταση στόχων ασφάλειας που αφήνουν επαρκές περιθώριο στις εθνικές αρχές υπεύθυνε για την ασφάλεια για να ευθυγραμμιστούν και να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές σύμφωνα όμως και με τις δικές τους εθνικές διατάξεις και επιταγές. Γι' αυτό στις προτάσεις μας έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο να εξασφαλίσουμε πως θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς μέσω ενός συστήματος peer review. Τι σημαίνει το peer review. Δεν σημαίνει έλεγχο και δεν σημαίνει και παρέμβαση στα δικαιώματα που διατηρούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές. Το peer review, η αξιολόγηση από από, ισότιμα, από ισότιμους εταίρους εξασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σε υψηλό επίπεδο, τις βέλτιστες πρακτικές και είναι ένας τρόπος για να εναρμονίσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται όλοι, δηλαδή με χρήση των βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο νομίζω αποτελεί κοινό μας στόχο. Για να απαντήσω σε μια παρατήρηση που έγινε για το κατά πόσο είναι πρόημη η πρόταση, το να μας ε, θεωρείται πρόημους μετά από δυόμιση χρόνια μετά την Φουκουσίμα και μετά τις πολλές εκθέσεις ε, που προέρχονται από την Ιαπωνία, κατά τη γνώμη μου είναι κάπως υπερβολικό. Η πρόταση, όπως σας είπα, συζητήθηκε εκτεμένα και συζητήθηκε και με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας που αποτελείται από επιστήμονες που προέρχονται από τις ρυθμιστικές αρχές για την πυρηνική ενέργεια, οι οποίοι μας πρότειναν και αυτό το σύστημα της θεματικής αξιολόγησης μέσω peer review. Θεωρούμε πως η χρονική στιγμή είναι η κατάλληλη, πως το σύστημα το οποίο εμείς παρουσιάζουμε είναι επίσης ορθό και για τη σύγκριση συμφερούντων και για το κατά πόσο εμείς θέλουμε να είμαστε ρυθμιστική αρχή για την πυρηνική ενέργεια, μια και αυτό ακούστηκε επίσης. Η απάντηση είναι πως δεν υπάρχει δεν έχουμε καμία φιλοδοξία να γίνουμε εμεί ο ρυθμιστής για την πυρηνική ενέργεια, γιατί αυτό θα έρχονταν σε αντίφαση με τις αρχές τι οποίε μόλι περιέγραψα και κυρίως με την αρχή της ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων για την ασφάλεια, όπως επίσης και με την αρχή της διαφάνειας στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Αυτό το οποίο προτείνουμε εμεί στο άρθρο το οποίο έχει να κάνει με την θεματική peer review, είναι αντίθετα να στήσουμε ένα στεναρό μηχανισμό και ένα στεναρό σφριγγυλό σύστημα λήψη αποφάσεων όταν, όπου στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συμφωνία για το πώς θα διεξαχθεί η θεματική peer review, θα ορίζει έναν τελικό λήπτη αποφάσεων που θα εξασφαλίζει πως κάθε έξι χρόνια θα γίνονται αυτές οι αξιολογήσεις. Αυτά επί της ουσίας Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο χρονικό προγραμματισμό και στην έγκριση αυτών των προτάσεων ε, μέσα σε τούτη τη θητεία και γι' αυτό χαιρετίζω ιδιαίτερα τα όσα μόλις μας δήλωσε η συγγήτρια. Δηλαδή, πως έχει προχωρήσει πολύ στην ε, προετοιμασία της γνωμοδότησης και ελπίζουμε και εμείς πως θα ακολουθήσουμε μια ταχεία ε, διαδικασία όπου και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα αποφασίσουν για την τύχη αυτού του φακέλου. Ναι, ευχαριστώ. Το λόγο έχει συγγήτρια. Είναι συντομία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου για τα σχόλια. Σύντομα τώρα, σχετικά με την πρόταση. που είναι βεβαιασμένη όπως είπαν κάποιοι. Όχι. Θεωρώ ότι όντως πρέπει να αντιδράσουμε υπεύθυνα και έγκαιρα. Και άλλωστε το Κοινοβούλιο ήταν πολύ πιο θετικό ήδη από το 2008 και 2009 για τη σχετική αναθεώρηση. Πριν να δράσει μάλιστα το Συμβούλιο. Θα ζητήσω τώρα από τους και οδησηγητές, μετά την πρωτοχρονιά, να συναντηθούμε, να συντάξουμε μαζί όσο γίνεται περισσότερες συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ την κυρία Τζόρνταν. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Αρχόλα. σε σχέση με την ε, γνωμοδότηση για τα δικαιώματα του αερίων του θερμοκηπίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περιλήφθηκε η ε, περιλήφθηκαν οι ενέργειες μεταφορές στο ETS από την αρχή και αντιμετώπισαν αμέσως οι χώρες μέλη μέτρα αντιπίνων λόγω της απόφασης εκείνης από τις τρίτες χώρες. Χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα και οι Ινδίες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τους δικούς μας κανόνες. Αυτά τα μέτρα αντιπίνων αποδυνάμωσαν πολύ την ανταγωνιστικότητα των αερογραμμών μας και το δυναμικό ανάπτυξής τους. Για αυτό τον λόγο πέρσι μετά από διεθνή πίεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να κάνει ορισμένα βήματα πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να προχωρήσει σε ένα πάγωμα του χρόνου έτσι ώστε να δημιουργηθεί θετικό κλίμα διαπραγματεύσεων για τον ε, Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας για τη Γενική Συνέλευσή του δηλαδή, η οποία διεξήχθη τον Οκτώβριο. Αυτό το stop the clock, το πάγωμα του χρόνου, αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν σόφρον επιλογή και βοήθησε τον οργανισμό πολιτικής αεροπορίας ΙΚΑΟ να σημειώσει σημαντική πρόοδο και τώρα συνάφθηκε συμφωνία για να ληφθούν μέτρα αγορακεντρικά για το 2016. Βέβαια, με την οδηγία αυτή τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι προχωρεί να δράσει μόνη της, προτείνοντας ένα airspace model, όπου όλες οι πτήσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εμπίπτουν στο σύστημα ε, εμπορίας των ε, εκπομπών και αυτό για τα έτη 2014 έως 2020. Η επιβολή όμως της κοινοτικής νομοθεσίας στις εταιρείες τρίτων χωρών πάλι δίνει αφορμή για πολλές επικρίσεις και αποτελεί κίνδυνο να ξαναδούμε τέτοιους εμπορικούς πολέμους και μέτρα αντιπίνων πριν, όπως πριν από το πάγωμα του χρόνου. Όλες οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης αντιτίθεται στην πρόταση αυτή γιατί γνωρίζουν ότι θα υποστούν ζημία. Το ίδιο ισχύει για την IATA, International Air Transport Association και Επίση για την Ένωση Ευρωπαϊκών Αερογραμμών. Και μεγάλος αριθμός χωρών μελών αντιτίθενται, διότι είναι προφανής η κίνδυνη. Και άλλωστε το κέρδος θα ήταν τόσο μικρό υπέρ του κλίματο. Σε σύγκριση με ένα συνολικό ETS, εδώ καλύπτονται μόνο 38% των εκπομπών, ενώ σύμφωνα με το σύστημα που προτείνω εγώ είναι, μόνο, είναι λίγο κάτω από 30%. Είναι πολύ μικρό λοιπόν το πρόσθετο αυτό κέρδος του 8%. Εγώ για μεγάλο διάστημα είχα την εντύπωση ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε μια παγκόσμια ε, συμφωνία υπέρ του κλίματος. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έμονη ιδέα με το δικό της πρόγραμμα και η στάση της προκαλεί δισταγμό απέναντι στους άλλους ενδιαφερομένους. Ειδικά για το ETS των ε, εναερίων μεταφορών, τους άκουσα να λένε εμείς ναι, να μειώσουμε τα εκπομπές ε, καυσαερίων, αλλά γιατί προσπαθεί με το, με το ζόρι να μας και να καταπιούμε το σύστημά της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ματαιοδοξία, ρωτώ εγώ. Πρόκειται για κάποιο είδους ε, πολιτική φιλοδοξία. Αυτά που ακούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την συμπεριφορά της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την στάση της δυστυχώς θέτουν σε κίνδυνο το θετικό κλίμα διαπραγματεύσεων το οποίο δημιουργήθηκε πρόσφατα με την Ένωση ε, Πολιτικής Αεροπορίας. Γι' αυτό προτείνω εγώ να συνεχιστεί αυτό το πάγωμα του χρόνου με το ETS μέχρι το 2016 και να μην, ε, να μην προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τίποτε στους διεθνείς μας εταίρους, γιατί θα ξαναγίνει η Γενική Συνέλευση του ΙΚΑΟ το 2016, όπου αναμένεται να συναυθεί διεθνή συμφωνία. Και για να υπάρξει πραγματική παγκόσμια ε, λύση, σε συμφωνία δηλαδή, πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την θετική κίνηση. Και μέσα εκεί μπορεί η Ένωση να δείξει ε, πρωτοπόρο ρόλο, αλλά με πιο ευφύ τρόπο. Τα σχέδια όμω τώρα της Κομισιόν θέτουν σε κίνδυνο τη διαδικασία του ΙΚΑΟ που ωστόσο μέχρι τώρα υπόσχονται πολλά και είναι το μόνο όργανο μέσα στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί διεθνή συμφωνία. Θα ήταν λοιπόν ματαιόδοξο και λάθος, ανόητο να επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που υποστηρίζεται ένας παγκόσμιος μηχανισμός και απ' έξω από την Ευρώπη. Για πρώτη φορά και από μεγάλη φορείς συμμετέχουν και αυτοί. Δεν πρέπει να μπλοκάρουμε να αναχαιτήσουμε αυτή την πρόοδο με δικές μας εσωτερικές δράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Κράμερ, παρακαλώ. Äh, Ευχαριστώ. Εγώ είμαι σκιώδης συγητής των φιλελευθέρων και ίσως να εξηγήσω κάπως πιο γλαφυρά το τι συμβαίνει. Εδώ και 6-7 χρόνια από ό,τι το, το έκανε η κυρία Κόρχολα. Ήμουν ε, τότε εγώ ε, ουσιώδης από την αρχή θέλησαν να μας βάλουν μέσα. Από την αρχή, από την πλευρά των τρίτων χωρών, όμως υπήρξε αντίδραση, διότι πρώτον αυτές θεώρησαν ότι δεν διαβουλευτήκαμε μαζί τους και δεύτερον αντιστάθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή έδειξε αμετακίνητη, δεν έλαβε υπόψη τις αντιδράσεις αυτές. Η κυρία Κόρχολα είπε προηγουμένως ότι το πάγωμα του χρόνου ήταν σωστό εγώ θα πω μάλιστα ότι ήταν μια υποχώρηση της τελευταίας στιγμής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε μια πολύ στεναρή διεθνή αντίσταση. Στην τελευταία συνέλευση του ΙΚΑΟ προ λίγων εβδομάδων καταλήξαμε σε μια πολύ ασυνήθιστη διαδικασία που δεν συμβαίνει συνήθως στον ΙΚΑΟ, δηλαδή σε μαχητική ψηφοφορία η οποία είχε ως αποτέλεσμα μοντέλα airspace, αέριου χώρου δηλαδή, να απορριφθούν καθαρά από τον ΙΚΑΟ ως επιλογή. Για μένα λοιπόν είναι απολύτως ακατανόητο τώρα, μετά από το απαραίτητο βήμα που έπρεπε να κάνουμε, να έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υποβάλει μοντέλο που είναι απόλυτα σαφές ότι πάλι και με αυτό δεν θα πρόκειται να πετύχουμε τίποτε περισσότερο παρά συγκρούσεις με τρίτες χώρες. Νομίζω ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να σεβαστούμε τη διαδικασία του ΙΚΑΟ που, ε, στην οποία με τόσο κόπο έχουν καταλήξει και τον οδικό αυτό χάρτη μέχρι το 2016. Ας δείξουμε επιτέλους επικοδομητική συμπεριφορά και ας μην προκαλέσουμε και πάλι. Για να το πω λοιπόν πολύ καθαρά, δεν είναι πλέον θέμα πολιτικής θέλησης, εάν θα έχουμε airspace approach για τις εκπομπές, είναι ζήτημα αποδοχής μιας διεθνής καταστάσεως η οποία έχει πλέον δημιουργηθεί. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε το δικαίωμα μας απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, όταν δεν συμφωνεί ο υπόλοιπο κόσμο. Διότι αλλιώ θα καταλήξουμε πάλι εκεί που είχαμε καταλήξει λίγο πριν από το πάγωμα του χρόνου. Δηλαδή είχαμε προκαλέσει συγκρούσει συμφερόντων και πραγματικέ συγκρούσει, διότι η Κίνα, αν θυμάστε, ακύρωσε παραγγελίε αεροσκαφών Airbus. Όλα αυτά ας τα λάβουμε υπόψη. Συμφωνώ με την κυρία Κόρχολα στην αξιολόγησή τη όταν λέει η ίδια ότι η κοπιώδη σε αυτή τη διαδικασία που περνά τώρα ο ΙΚΑΟ και περνάμε και εμείς δηλαδή, υπονομεύεται και θα υπονομηθεί, θα και ίσως θα ανατραπεί εν τέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πολλές χώρες του κόσμου θα πούν «Α, να τι πάλι οι Ευρωπαίοι έρχονται με τις ιδέες τους που κανένας άλλος δεν θέλει να αποδεχθεί στον κόσμο και με τον τρόπο αυτό κινδυνεύουν να ανατρέψουν τον κάπως ασταθή συμβιβασμό που μπορέσαμε τον οποίο μπορέσαμε να καταλήξουμε. Για μένα είναι σαφές ότι πρέπει τουλάχιστον να συνεχίσουμε το πάγωμα του χρόνου τουλάχιστον μέχρι το 2016 ίσως και περισσότερο από το stop the clock ακόμα καλύτερα να αφήσουμε εντελώς απ' έξω τις αεροπορικές γραμμές τις αεροπορικές μεταφορές από το ETS γιατί δεν προσφέρει, δεν είναι σχεδόν κανένα ωφέλιμα και το μόνο που αποτελεί είναι μειονέκτημα ανταγωνισμού για τις ε, ευρωπαϊκές αεροπορικέ εταιρείε Είναι μια απλή ανακατανομή χρήματο, η οποία για το κλίμα δεν αποφέρει τίποτα το θετικό. με τον χρόνο, λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Τζόρνταν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ συνήθως συμφωνώ με τα όσα λέει η συνάδελφος κυρία Κόρχολα, αλλά σήμερα δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει αν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζαμε το 2008 ότι ως κοινωνία θα μειώναμε τις εκπομπές, τότε επειδή ακριβώς λάβαμε αυτή την απόφαση θα πρέπει όλοι οι κλάδοι να μοιραστούν αυτή την προσπάθεια. Οι άλλοι κλάδοι επίσης πρέπει να έχουν αναλάβει ένα μεγάλο μέρος αυτού του ε, βάρους και οι αερομεταφορές δεν το έχουν κάνει. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει αυτή την αρμοδιότητα και να ορίζει μέτρα στη δική της ε, επικράτεια. Ποτέ δεν συμφώνησα με αυτό το πάγωμα του χρόνου, το stop the clock. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια ήττα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκανε παραχωρήσεις για τρίτες χώρες. Στη Βαρσοβία πήγα στην ε, σχετική διάσκεψη και πρέπει να σας πω πως συναντήθηκα με ε, εκπροσώπους του ΙΚΑΟ, μας εξήγησαν ποια είναι τα σχέδιά τους. Το γεγονός πως θέλουν να καταλήξουν συμφωνία μέχρι το 2016 και μετά να μειώσουν τις εκπομπές μετά από το 2020, το αντιμετωπίζουμε αρκετό σκεπτικισμό, γιατί το 2001 ο ΙΚΑΟ είχε αναλάβει τη δέσμευση να ετοιμάσει μια συμφωνία για το θέμα αυτό και ακόμα δεν έχει καταφέρει τίποτα. Ξέρουμε πως η συμφωνία του Κιώτο δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Αν δείτε λοιπόν το τι συμβαίνει σε επίπεδο ΙΚΑΟ, είναι μάλλον χειρότερη η κατάσταση από αυτά που έχουμε στην ε, σύμβαση, στη συμφωνία του Κιώτο. Επίσης, οι εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις προσδοκίες μας μέχρι το 2020. Γιατί μέχρι τότε οι άλλοι κλάδοι της Ευρώπης θα έχουν μειώσει τις εκπομπές τους κατά 20% και για τον λόγο αυτό δεν μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα μόλις άκουσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ πραγματικά έχουμε ενώπιον μας ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και οφείλεται και σε μία υπόθεση της Κομισιόν ότι θα μπορούσε να έχει τόση κυριαρχία που θα ζητούσε από όλο τον κόσμο να την ακολουθήσει. Εγώ νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε βέβαια σε μια τέτοια κατάσταση. Οι διαπραγματεύσεις στη Βαρσοβία ουσιαστικά πέτυχαν και επομένως εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο παρουσίασης της συμφωνίας αυτής. Ουσιαστικά θα πρέπει να βασίζεται πολύ περισσότερο σε μία δικαιοσύνη και ισοκατανομή σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Επίσης, νομίζω ότι υπάρχει και αναγκαιότητα να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ανάγκη ανάληψης δράσης. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Οργανισμός ε, Πολιτικής Αεροπορίας είναι το πλέον κατάλληλο βήμα όπου θα πρέπει να γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Και εγώ νομίζω ότι Κάτι που θα μπορούσε να γίνει σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να είναι μία πρόταση που να μην είναι ένας μηχανισμός αγοράς, αλλά ένας φόρος ε, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί εγώ νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να στοχεύσουμε το να πετύχουμε μια συμφωνία δυνάμει της ε, σοβαρότητας, της βαρύτητας του ζητήματος και θα μπορούσε αυτή να είναι μια αρχή που θα μπορούσε και να εξελιχθεί προς μια καθολική παγκόσμια συμφωνία όταν καταρθώσουμε να την πετύχουμε. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να δω κάποιες διαπραγματεύσεις με τον Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας στη βάση μιας ε, αποδοχής ενός ε, φόρου για τα καύσιμα, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε ήδη να δώσει κάποια απαραίτητα έσοδα για να προβούμε σε κάποιες επίγουσες ε, παρεμβάσεις στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής και επίσης να αναγνωρίσουμε ότι οι χώρες που έχουν μεγάλο απόθεμα άνθρακα στα τροπικά δάση, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ήδη σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναγνωρίσουμε στις χώρες αυτές ότι ουσιαστικά ένα τροπικό δάσος που την χάνει της κατάλληλης εποπτείας ωφελεί τους πάντες. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο αφετηρίας και με κάποια μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις με τις οποίες θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη συμφωνία. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το θέμα αυτό. Όμως, με συντομία, αυτό στο οποίο αναφέρομαι είναι η κλιματική δικαιοσύνη. Δηλαδή, μία πρόταση που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και μία απάντηση στη δήλωση του Μπαλίου. Υπάρχει αναγκαιότητα να αναλυφθούν πολιτικές δεσμεύσεις κατόπιν της διακήρυξης του Μπαλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέρκης που είναι σκιώδης, παρακαλώ. Κυρία, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Νομίζω ότι η θέση της εισηγητρής επίσης είναι σαφής. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω μια κάπως αποκλίνουσα άποψη και βασίζομαι και στις παρελθούσες προθέσεις μας. Νομίζω ότι η εισηγήτρια πιστεύει υπερβολικά κάπως στον ΙΚΑΟ, στον Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν έλαβε ο Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας ε, μια δεσμευτική συμφωνία εγώ δεν έχω δει καμία δεσμευτική συμφωνία ακόμη και πρέπει, ναι, να συγχαρώ τον κλάδο, τον τομέα, με πολύ καλές προθέσεις, όμως οι προθέσεις δεν είναι δεσμευτικές. Η συμφωνία του ΙΚΑΟ, λοιπόν, καλεί μόνο για να ληφθεί κάποια δράση, για να υιοθετηθούν κάποια παγκόσμια μέτρα σε 7 χρόνια. Γι' αυτή η διαδικασία ξεκινήσει το 2016. Βέβαια, είναι, εξακολουθεί να μην είναι ξεκάθαρη η πρόοδος που έχει γίνει. Έτσι λοιπόν, ε, επομένως, ε, μόνο μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ε, όλη διαδικασία και νομίζω ότι πρέπει να την προωθήσουμε, να την οθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο σκοντας πίσω στον ΙΚΑΟ να φτάσει σε αυτή τη συμφωνία. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι μία προσέγγιση ενερίου χώρου είναι εδώ που πρέπει να ακολουθήσουμε από το 2014 στο 2016. Τρεις λόγοι. Γι' αυτό είναι καλύτερο για το περιβάλλον, καταρχήν και αυτό ήταν ο κύριο στόχο. Η προσέγγιση αυτή συμπεριλαμβάνει το 40% των εκπομπών σε σύγκριση με τον αρχικό κανονισμό ETS ε και το πάγωμα του χρόνου ε, θα μα οδηγούσε μόνο στο 20%. Δεύτερο λόγο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υποχωρήσει σε πίεση χωρών όπω η Κίνα το έχουμε δει αυτό σε όλες τις ε, διασκέψεις των μερών ε, και είδαμε ότι η παγκόσμια πολιτική για το κλίμα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως ε, Βέβαια, αν έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους, ε, θα πρέπει να κάνουμε και μία αξιολόγηση και να δούμε αν μας ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Πρέπει να δούμε και πίσω μας τι συμβαίνει. Όμως, αν υπάρχει πρόθεση παγκοσμίω ε, να καταλήξουμε συμφωνία, δεν πρέπει να υποχωρήσουμε σε πίεση χωρών όπως η Κίνα και το πάγωμα του χρόνου θα θεωρείται ως παράδοση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να διατηρήσουμε τη φιλοδοξία μας μέχρι το τέλος. Και τρίτον, εδώ δίνονται κάποια κίνητρα να πετύχει τη συμφωνία μέχρι το 2016. Μετά το 2016 η διάσκεψη του ΙΚΕΟ θα έπρεπε να υποβα... η Κομισιόν συγγνώμη, θα έπρεπε να υποβάλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε σχέση με τον πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί για την εφαρμογή ενός μηχανισμού αγορακεντρικού μέχρι το 2020. Εγώ θα καταθέσω κάποιες ε, τροπολογίες που θα λένε ότι αυτή η παρέκκληση πρέπει να ισχύει μόνο μέχρι το 2016. Και τέλος θέλω να τονίσω τη σημασία των απαιτήσεων παρακολούθησης γιατί οι αερομεταφορείς έχουν πει ότι τους, έχουν έχει βοηθήσει η παρακολούθηση και αν ε, τελικά αφαιρέσουμε ε, αυτές τις απαιτήσει, θα στείλουμε ένα λανθασμένο μήνυμα στους αερομεταφορείς. Ευχαριστώ πάντως την εισηγήτρια και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας ε, και φυσικά θα παρουσιάσω και κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Ράμστορ, παρακαλώ. Thank you very much for... Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία αυτή ε, να τοποθετηθώ κι εγώ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η περιβαλλοντική κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν με τολμηρές τεχνολογικές αλλαγές και κοινωνικές προσαρμογές. Σε ολόκληρο τον κόσμο έχουμε πάνω 700 εκατομμύρια αυτοκίνητα και εκατοντάδες χιλιάδες αεροσκάφη. Αυτό μπορώ να σας πω λοιπόν είναι ότι υπάρχουν σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες ήδη διαθέσιμες. Στη χώρα μου για παράδειγμα διαθέτουμε την ευρεσιτεχνία για μείωση εκπομπών στα οχήματα που μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε όχημα ανεξαρτήτως της ηλικία του στη βάση ενός εξοπλισμού που μειώνει τις εκπομπές κατά 70%. Πρόκειται για ένα φίλτρο και πυκνοτή ταυτόχρονα που όπως είπα μειώνει τις Έχουμε πει ότι το 70% μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αεροσκάφη και στην παραγωγή ενέργειας. Το πρόβλημα είναι όμως ότι είναι πολύ φθηνό. Για την παραγωγή του εξοπλισμού αυτού δεν χρειάζεται παραπάνω από 100 κορώνε, δηλαδή 5 δολάρια. Αντί για 60.000 κορώνε που κοστίζει ένα καταλήτη. Είναι πολύ ακριβότερο ο καταλήτη, αλλά βεβαίω ήδη τον έχει εισαγάγει η αυτοκινητοβιομηχανία και διαθέτει σημαντικό λόμπι το οποίο ανθίσταται σε κάθε καινοτομία. Άλλη καινοτομία που θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση του κλίματος είναι ευρεσιτεχνία για την τσιμεντοβιομηχανία. Πολύ πρόσφατη ευρεσιτεχνία ενός μηνός ηλικίας όπου με την ε, συμπερίληψη κεραμικών υλικών η εφεύρεση αυτή μειώνει την χρήση ενέργειας και πρώτων υλών στην τσιμεντοβιομηχανία η οποία είναι ιδιαίτερα εντατική ενέργειας αλλά και χρησιμοποιεί και πολλές πρώτες ύλες πάλι κατά 70%. Το πρόβλημα λοιπόν που βλέπω εγώ είναι ότι οι κανόνες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν το εμπόδιο. για να προχωρήσει η καινοτομία και η τεχνολογία. Οφείλω να πω ότι στην έκθεση που συνέταξε η συνάδελφός μας Κόρχολα εκτίμησα ιδιαίτερα όχι μόνο το επίπεδο του προβληματισμού της αλλά και την προσωπική της ταύτιση με το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Grazie. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που κάνετε. Νομίζω πως όντως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά περίπλοκη πολιτική ε, συγκυρία γιατί Βεβαίως οι προτάσεις αυτές έχουν γίνει δεκτές με πολλά σχόλια υπέρ και κατά. Δεν έχουμε και την συναπόφαση που μας επιτρέπει ε, να συνεχίσουμε με την με έχουμε και τη συναπόφαση η οποία μας επιτρέπει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου ε, να στήσουμε ένα νομικό μέσο ε, διαφορετικά ε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα παρά να μείνουμε στα σημερινά πλαίσια. Έχοντας πάει στην συνέλευση του ΙΚΑΟ και έχοντας δει τι, πρόοδο τι πρόοδος έχει σημειωθεί ε, σημειωθεί εκεί πιστεύω πως το να εφαρμόσουμε τα όσα έχουμε στη συμφωνία θα ήταν μια πρόκληση. Όμως χρειάζεται να συμπεριλάμουμε και τον ΙΚΑΟ ε, γιατί θα αποτελέσει το βασικό εφαλτήρα για να έχει παγκόσμια διάσταση ή οποιαδήποτε ε, προσπάθεια η οποία θα κάνουμε και είναι δύσκολο να προβλέψουμε ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή μιας διαφορετικής προσέγγισης από αυτήν την οποία προκρίνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική μας πρόταση έχει σκοπό να διασκεδάσει τις ανησυχίες των ε, ε, εταίρων μας για ε, καταρχήν την εδαφική κάλυψη των όσων έχουμε θεσμοθετήσει. Η πρότασή μας συμπεριλαμβάνει όλους τους ε, αερομεταφορείς ανεξάρτητα από την καταγωγή τους αλλά μόνο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αποκλείουμε ε, ε, κανέναν αλλά δεν μπορούν οι αερομεταφορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιούνται με διαφορετικούς κανόνες από τους Ευρωπαίους στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ξέρετε πως οι πολυεθνικές πάντα σέβονται ε, τον ε, νόμο του τόπου. Εάν δεν σεβαστεί κανείς τον νόμο του τόπου, δεν μπορεί να ασκεί με σωστό τρόπο αυτή την ε, πολυεθνική επιχειρηματική δράση. Άρα λοιπόν για τις αερομεταφορές ξέρω ότι χρειάζεται μια σφαιρική προσπάθεια αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ο κλάδος αυτός να εξαιρεθεί μια και οι εκπομπές εκεί αυξάνονται συνέχεια. Επίσης, ε, κατανοώ ε, το ψήφισμα του ΙΚΑΟ και θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μας και με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να εξηγήσουμε πώς η προσέγγιση μας ευθυγραμμίζεται με τις συζητήσεις που έγιναν ε, στον ΙΚΑΟ. Νομίζω πως η πρότασή μας έχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ των ιδιάζοντων συνθήκων ε, με τον κανόνα του ελαχίστου για κάποια θέματα το de minimis και παράλληλα εξασφαλίζοντα ισότιμε συνθήκε παιχνιδιού για όλου. Οι ερμηνείε του ψηφίματο του ΙΚΑΟ που οδηγούν στη σκέψη πω η πρόοδο αποτελεί εμπόδιο για την ε, ταχεία δράση και όπου περικόπτει τα, τα κυριαρχικά δικαιώματα των διαφόρων εμπλεκομένων να ε, λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα είναι τουλάχιστον αφελής. Αυτή η ταχεία δράση δημιουργεί ακριβώς το δυναμικό που θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε τα μέτρα ε, υπέρ των οποίων έχουμε όλοι δεσμευτεί. Για την γενική αποδοχή ε, και συμμόρφωση, πρέπει να σας πω ότι το 98% των εκπομπών διοξιδίου που καλύφθηκαν με το καθεστώς του 2012 είναι σε απόλυτη συμμόρφωση και αυτό σημαίνει ότι και οι αερομεταφορείς από τη ΣΥΠΑ έχουν συμβιβαστεί με τη δική μας νομοθεσία. Αν πρόκειται λοιπόν να εξαιρέσουμε κάποιους μεταφορείς οι οποίοι δεν επέλεξαν να συμμορφωθούν, θα έχουμε πρόβλημα διακρίσεων, άρα λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει η κοινοτική νομοθεσία και στο μέλλον. Πρέπει να μας πείσετε εάν υπάρχει προσθέμενη αξία σε άλλη προσέγγιση από τη δική μας. Και ελπίζουμε να παραμείνουμε όλοι στρατευμένοι υπέρ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ε, συναπόφασης ε, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει και να συνεχίσουμε με την εφαρμογή του καθεστώτος αυτού. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, είμαι πεπισμένη από τα μόλις είπε η Κομισιόν, μπορώ να πω. Εγώ διάβασα προσεκτικά το αιτιολογικό υπόμνημα και με εκπλήσει αυτή η λογική. Λέγεται το εξής αναφέρεται στον ΙΚΑΟ και στην επιτυχία του ΙΚΑΟ στο καλό της συνεδρίας του Σεπτέμβριο και συνεχίζει ως απάντηση στην πρόοδο αυτή και για να προωθήσουμε πλέον την ορμή προς την επιτυχή λήψη παγκοσμίων αγορακεντρικών μέσων θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροπολογίες κτλ. Πραγματικά με εκπλήσει αυτό γιατί γενικά το feedback ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή αυτό που προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πολύ από το να δημιουργήσει επικοδομητικό κλίμα ή να προωθήσει την περαιτέρω όθηση. Σας ευχαριστώ κύριε Κράμερ για το feedback. Χαίρομαι που μπορούμε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό τώρα για την κυρία Τζόρνταν. Θέλω να σας ρωτήσω, αναρωτιέμαι μήπως έγινε κάποια παρεξήγηση. Γιατί εγώ νόμιζα ότι εσείς ε, αναφερθήκατε στο ότι θέλετε να συνεχιστεί το Ευρωπαϊκό ETS, όμως θα συνεχιστεί αυτό. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών για την Ευρωπαϊκή θα συνεχιστεί εντό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή η Ευρώπη θα ακολουθήσει τον τρόπο που έχει επιλέξει. Τώρα εδώ μιλάμε για την επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας και γι' αυτό δεν θα πρέπει να ξαναγκάσουμε τους υπολείπους. Γιατί θα χαλάσει η καλή ατμόσφαιρα, το καλό κλίμα. Έτσι λοιπόν, αν είπατε ότι θα πρέπει να προσέξουμε τι συμβαίνει με την αεροπορία, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για ότι θα λάβει και ένα μέρος της μείωσης, σχόλιο εκτός μικροφώνου, ναι, ναι, αλλά η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. 38% έναντι του 30%. Και αν λόγω αυτού του 8% θέσουμε σε κίνδυνο την επίτευξη της Παγκοσμίας Συμφωνίας, νομίζω ότι είναι πολύ ανησυχητικό αυτό και για την κυρία Μέρκης. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δεσμευτική συμφωνία στον ΙΚΑΟ. και θα πρέπει να λάβει χώρα αυτό το 2016. Και ένα γενικό σχόλιο. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Το έχω ακούσει πολλάκις. Όμως θέλω να ζητήσω από τους συναδελφούς να σκεφτούν τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Μπορούμε τις μονομερείς δράσεις να τις αποκαλούμε φιλόδοξες. Αν ε, τώρα θέσουμε σε κίνδυνο, διακυβεύσουμε αυτή την ε, παγκόσμια συμφωνία με την ε, συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν είμαστε φιλόδοξοι, γιατί δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Και το τι συμβαίνει σήμερα με το ETS μας δίνει κάποια ανησυχητικά παραδείγματα, γιατί έχουμε δει ήδη ότι κατά τη διάρκεια αυτών των μονομερών ακριβών συστημάτων εμπορίας εκπομπών η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εκπομπές της, αν λάβουμε υπόψη το σύνολο των εκπομπών και κατανοούμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εισαγόμενες εκπομπές και αν δούμε όχι μόνο την παραγωγή αλλά και την κατανάλωση θα δούμε ότι εισάγουμε λένε και περισσότερες εκπομπές. Και σύμφωνα με τις διεθνείς εμπορικές στατιστικές μπορούμε να δούμε ότι από τη στιγμή που λάβαμε μέτρα για το κλίμα, αυξήσαμε το σύνολο των εκπομπών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μονομερούς πολιτικής. Επομένως, εξακολουθώ να είμαι ιδιαίτερα επικριτική απέναντι σε μονομερείς επιλογές. Όμως, σας είπα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική, αλλά δεν είναι σοφό αν αυτό χαλάσει το κλίμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι την 5η και 9 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή στις 10 και 4 Έχουμε μία κοινή συνεδρίαση επιτροπών με το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 21ο αιώνα. Επίσης, να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι απόψε, από τις 6 και μετά έχουμε ένα κοκτέιλ, μια δεξίωση για τα Χριστούγεννα. Έτσι λοιπόν, σας καλώ όλους να παρευρεθείτε. Σας ευχαριστώ.